Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήλθατε. Ο πρόεδρος έχει κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή του και γι' αυτό μου ζήτησε να σας βοηθήσω να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση στο σημείο 11. Καλωσορίζουμε τον κύριο Τιμόφσκι, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις αξιολογήσεις ε, ex Εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Έχετε το λόγο κύριε Τιμόφσκι για 15 λεπτά. Για μια ακόμη φορά σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στην Αγγλική. Ξεκινώντας θα ήθελα να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ γιατί πριν 12 χρόνια ακριβώς ξεκίνησα να δουλεύω στην γραμματεία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ήμουν εδώ όταν έγινε δεκτή η οδηγία για τη διαμεσολάβηση Ήμουν υπεύθυνο τότε μεταξύ άλλων και για την οδηγία ADR. Έχω εμπλακεί εν μέρη λοιπόν με πολλά από τα θέματα αυτά, τα οποία πρόσφατα κλήθηκα να μελετήσω σε βάθος. Η μονάδα μας για την αξιολόγηση των συνεπειών ex post και έχω μαζί μου και τον Ρούφας Κουιντάνα που είναι ο γραμματέας της ομάδας αυτής ασχολείται με τα θέματα των εκθέσεων εφαρμογής. Βλέπετε μπροστά σας τρία παραδείγματα. Το πρώτο σας είναι ιδιαίτερα γνωστό, αυτό που είναι στο δεξιό τμήμα. Κάνουμε αξιολογήσεις είτε στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου είτε εξωτερικές, βοηθώντας να κατανοήσουμε το επίπεδο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου Στην περίπτωση της οδηγίας του 2008 ε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια λοιπόν από τότε που έγινε δεκτή και μεταφέρθηκε στις εθνικές νομοθεσίες και αυτό μας επιτρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Το έγγραφο που σας έχει διανεμηθεί πριν λίγες ημέρες και έχετε νομίζω μπροστά σας τώρα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια που γίνεται με την ε, νέα έκθεση. Το Νοέμβριο του 2016 κάποιοι εμπειρογνώμονες εξέτασαν το θέμα της εφαρμογής της συγκεκριμένης πράξης από τη δική του σκοπιά. Στο τέλος έχετε ένα πίνακα ο οποίος δείχνει όλες τις χώρες, ακόμα και την Δανία που έχει κάνει opt-out από την οδηγία, δείχνοντας πού ακριβώς βρίσκεται η κατάσταση και πώς εφαρμόζεται η συγκεκριμένη οδηγία. Κάποια στιγμή είχαμε πει ότι θα χρησιμοποιούσαμε το πράσινο και το κόκκινο όπως λέγαμε για να δούμε πώς πάει η εξέλιξη και είδαμε με χαρά ότι όπως θα σας πω και αργότερα το μοναδικό χρώμα ήταν το πράσινο, υπήρχε πράσινο φως. Ε, ναι μεν λοιπόν ο πίνακας είναι πραγματικά ασπρόμαυρος, αλλά ε, γενικά μπορούμε να τον κρίνουμε σαν θετικό. Ε, θα δούμε σε ποιο βαθμό είμαστε κοντά στους αρχικούς στόχους, θα δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και να δούμε αν έχουν γίνει σεβαστοί οι στόχοι αυτοί. Όπως είπα εμείς κάνουμε μελέτες και αναλύσεις και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου και ζητάμε και εξωτερικές γνώμες και σε σχέση με την αρχική πράξη και το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ε, εγώ θα συνεχίσω την παρουσίασή μου όχι υποχρεωτικά με την αρχιτεκτονική του εγγράφου που σας είχε διανεμηθεί. Καταρχάς, βασικά νομικά πλαίσια, περιορισμός εμβέλειας και ε, οριακές καταστάσεις περιπτώσεις. Νομίζω ότι η νομική βάση επέτρεψε στην οδηγία αυτή να λειτουργήσει σε διασυνοριακές υποθέσεις. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη είχαν την δυνατότητα να ορίσουν την εμβέλεια και το έκαναν αυτό. Οι στόχοι της οδηγίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 1. Όταν εξετάζει κανείς, βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πολλοί στόχοι, όπως η διευκόλυνση πρόσβασης, διευκόλυνση της επίλυσης διαφορών και ισορροπημένη σχέση. Αξίζει να δει κανείς και το έβδομο τίτλο όπου στην ουσία ε, τίθεται ο όρος νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα είναι απαραίτητο για ένα προβλέψιμο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας. Αυτοί οι δύο όροι θα έλεγα, η ισορροπία από τη μία και προβλέψιμο από την άλλη δεν ορίζονται. Ε, κανονικά θα έπρεπε, αλλά παρόλα αυτά κάθε κράτος μέλος εξετάζει και ορίζει την προβλεψιμότητα και την ισορροπία με τον δικό του τρόπο και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Τα στοιχεία στους πίνακες μεταφοράς δείχνουν ότι χρησιμοποιούμε ένα benchmark τριετές ανεξαρτήτως αν είναι χρήσιμο να προσπαθήσει κανείς να αξιολογεί νωρίτερα, ε, κάποια στοιχεία τα οποία δεν εξετάζονται σε βάθος στη συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι περιλαμβάνονται δύο βασικές προτάσεις δεν ήταν αναμενόμενο από τα κράτη-μέλη να την μεταφέρουν κατά γράμμα, κάποιες το έκαναν, κάποιες όχι. Και ακόμα και αν στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην έκθεση της Επιτροπής που κυκλοφόρησε αργότερα αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη δεν επαναλαμβάνουν τους ορισμούς αυτούς όπως χρησιμοποιούνται στην οδηγία, Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει δημιουργήσει θέματα στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ρητρών. Uh, Τα κράτη-μέλη έχουν αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο το θέμα του αν οι δικαστές είναι οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές διαιτητές σε ορισμένες χώρες ε, βέβαια εξαιρείται απολύτως η δυνατότητα αυτή, σε άλλες ε, τίθεται το θέμα. Η οδηγία δεν το καθορίζει αυτό και περιλαμβάνει ε, μία φράση μάλιστα η οποία λέγει ότι δεν καλύπτεται η περίπτωση των δικαστών που εμπλέκονται στο να προσπαθήσουν να καταστήσουν τα μέρη, τα αντιτιθέμενα μέρη, πιο ικανά αν θέλετε ε, να αναζητήσουν μια αρρύθμιση, μια συμφωνία. Σε κάποιες χώρες έχουν γίνει και περαιτέρω βήματα και αυτό έχει οδηγήσει σε μια ποικιλία λύσεων για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαμεσολάβηση και πώς μπορεί κανείς ε, να χρησιμοποιήσει τη διαμεσολάβηση σαν μια εύκολη λύση για να προωθηθεί η υπόθεση. Αναφέρθηκα στην ισορροπία, αναφέρθηκα στην προβλεψιμότητα, σε ορισμένες από τις μελέτες τις οποίες έχουμε, φαίνεται ότι χώρες, κάποιες χώρες προσπαθούν να βρουν κάποια εφικτά benchmarks, δηλαδή ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται από την δυνατότητα της διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη το θέμα του κόστους και βλέπουμε ποσοστά όπως το 50%. Είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό να επιλεγεί ένα τέτοιο ποσοστό γιατί σε ορισμένες χώρες το 25% επιτυχίας ήδη ε, βελτιώνει την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στη δικαστική επίλυση. Ε, σε άλλες ε, το θέμα της διαμεσολάβησης είναι πολύ κοινό, οπότε ένα 75% ήδη αφήνει χώρο θα έλεγα βελτίωσης. Πριν συνεχίσω τώρα στις υποχρεώσεις οι οποίες προέρχονται από τα δικονομικά, ε, θα ήθελα να σας δείξω το τι έχουμε βρει εμείς σε σχέση με την ποιότητα ε, των διαδικασιών που ακολουθούνται. Είναι σαφές ότι οι προθέσεις είναι καλές και οι προθέσεις αυτές αντιμελέτες τις οποίες έχουμε κάνει και βλέπουμε πως η διαμεσολάβηση έχει εξελιχθεί στις διάφορες χώρες. Βασικός στόχος είναι να βρεθεί μια λύση η οποία να είναι ταχεία και υποβοηθητική της στήρισης των καλών σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες πλευρές και αυτό να φαίνεται και στα πλαίσια των συμβατικών διαδικασιών. Είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες όπου υπάρχουν απόψεις αντίθετες, αλλά κάθε χώρα μέλος ε, παραδοσιακά έχει ε, αρχές, έχει δικαστικές αρχές, διοικητικές αρχές που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Αν λοιπόν τα μέρη ενδιαφέρονται για την διαμεσολάβηση, ε, τότε μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι πολλές από τις διαδικασίες οι οποίες κανονικά θα έδιναν εγγυήσει ότι επιβάλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτώνται από την καλή βούληση, καλή θέληση των εμπλεκομένων. Και αν κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για διαμεσολάβηση. Αυτή η εθελοντική, αν θέλετε, πλευρά είναι κάτι το οποίο φαίνεται σε πάρα πολλές χώρες στις οποίες ενθαρρύνεται ε, η προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. Η οδηγία αφήνει ε, ελεύθερες τις χώρες να αποφασίζουν αν είναι υποχρεωτικός αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς. Και κάποιες από τις χώρες έχουν χρησιμοποιήσει την δυνατότητα αυτή. Είναι λοιπόν εθελοντική η χρήση, αλλά μπορούν τα κράτη αν θέλουν να επιβάλλουν τον κώδικα. Υπάρχει επίσης και η τάση αναφορά στον, στον ευρωπαϊκό κώδικα, αυτός δημιουργήθηκε τέσσερα χρόνια πριν από την υιοθέτηση της οδηγίας. Η οδηγία ουσιαστικά ήταν ένα περαιτέρω βήμα στα πλαίσια της εναρμόνισης των διαφορετικών πρακτικών και μεθόδων. Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους διασφάλισης της ποιότητας. Πάρα πολύ συχνά συνδέεται με τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να περνούν μέσα από διαδικασία καταγραφής ή και διαδικασία πιστοποίησης. Αυτή τη στιγμή υπάρξει μια συμφωνία για διαμεσολάβηση, τότε δημιουργείται η υποχρέωση σεβασμού αυτού του κώδικα συμπεριφοράς. Και στα θέματα της κατάρτισης τα μέσα ενημέρωσης αφαιρούνται από τον κατάλογο εφόσον δεν συνεχίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία κατάρτισης. Υπάρχουν μορφές στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπαίδευση των δικαστών σε θέματα διαμεσολάβησης. Ενθυμίστε ίσως την Diane Wallace, η οποία είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό ιδιαίτερο στο Κοινοβούλιο. Και επίσης και κάποιοι εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν ότι ανεξαρτήτως της υψηλής ποιότητας του κώδικα αυτού και ανεξαρτήτως των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι διαδικασίες στις διάφορες χώρες, η διαμεσολάβηση δεν θα χρησιμοποιείται εφόσον οι πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξή της. Ως εκ τούτου λοιπόν οι δυνατότητες που υπάρχουν δεν ικανοποιούν πλήρως τους τις υπηρεσίες αυτές. Υπάρχει μια ενθάρρυνση της συγκεκριμένης οδηγίας για τη διάδοση της ενημέρωσης, της πληροφορίας μάλλον, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς μπορεί να γίνει η ενημερωτική εκστρατεία με ε, δελτία τα οποία αφήνονται στα δικαστήρια, με σεμινάρια, με συναντήσεις. Υπάρχουν κίνητρα λοιπόν και τα κίνητρα αυτά αφαίνονται και στην επόμενη διαφάνεια. Σε όλα αυτά τα στοιχεία που άπτονται της ποιότητας εφαρμογής της οδηγίας, η φράση που λέγει ότι οι χώρες αποφασίζουν για τα κατάλληλα μέτρα, στην ουσία είναι μια οδηγία πλαίσιο με ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα που αφήνει πραγματικά πολλή ελευθερία στα κράτη-μέλη να πάρουν αποφάσεις. Αυτό δεν είναι κακό, είναι μια οδηγία παλαιού τύπου θα λέγαμε, παλαιού ρυθμού. Έχουν υπάρξει αλλαγές, οι αλλαγές όμως επέρχονται στις διάφορες χώρες με διάφορες ε, ταχύτητες. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αν θέλετε ένα τρόπο ο οποίος δεν θα είναι ο κατάλληλος για όλες ε, τις χώρες. Και ε, ήδη όταν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό στο παρελθόν είχα πει ότι θα πρέπει εμείς να ενθαρρύνουμε την διαμεσολάβηση αυτή στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει εναρμόνιση σε όλες τις καταστάσεις και σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, προτείνεται η δημιουργία νέων επιπέδων, και εδώ η οδηγία ADR όπως ακριβώς έγινε δεκτή και με την δική σας εμπλοκή γιατί η εμπλοκή ακριβώς είχε ζητήσει τη διεύρυνση της δυνατότητας εφαρμογής της. Έγινε τελικά δεκτή το 2013, λειτουργεί πλήρως σήμερα και μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εφαρμόζεται η οδηγία αυτή, έχουμε στοιχεία λεπτομέρειας, έχουμε ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν ακριβώς ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορές και αναφορές για τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις καταναλωτικών θεμάτων ε, και αυτό στο μέλλον θα μας επιτρέψει ανάλογα με τα στοιχεία που έχουμε να κάνουμε και τροποποιήσεις στη συγκεκριμένη οδηγία Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία τα οποία μεταφέρονται στα, στην εθνική νομοθετική, αν θέλετε, αρχιτεκτονική. Το πρώτο δεν είναι ακριβώς υποχρεωτικό βέβαια. Οι χώρες μέλη καλούν προς ενημέρωση. Ε, κάποιες ε, χώρες ε, μπορεί να θεωρούν ότι είναι υποχρεωτική η προσφυγή στην διαμεσολάβηση μετά από ενημερώσεις τέτοιου τύπου αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις. Να σας δώσω τρία, τρεις, Σαν παράδειγμα, οικογενειακό δίκαιο στην Κροατία, κυδαιμονία παιδιών στην Αυστρία και στην Ουγγαρία και άλλοι τομείς πολύ συγκεκριμένοι και πολύ περιορισμένοι, όπου η διαμεσολάβηση έχει πλέον καταστεί υποχρεωτική. Στην Ιταλία, σαν παράδειγμα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η διαμεσολάβηση μετά από κυβερνητικό διάταγμα προεβλέπεται ότι για να ελαφρυνθεί το δικαστικό σύστημα ε, έπρεπε να είναι υποχρεωτική η προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Αυτό λειτουργήσε, διευκόλυνε χρονικά, αλλά μετά για διαδικαστικούς λόγους δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται. Πάντως για να κλείνω την παρουσίασή μου, μπορεί να δοθούν και άλλα κίνητρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της ενθαρρύνει την χρήση των κινήτρων αυτών, κίνητρα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν με θετικό τρόπο έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάσουν την διαμεσολάβηση. Δεν το καθιστά ε, υποχρεωτικό βέβαια, αλλά μιας και μπορεί να είναι και φθηνότερη η διαδικασία και οι εμπλεκόμενες πλευρές θα δοκιμάσουν να τη χρησιμοποιήσουν. Μία απόπειρα διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση βέβαια να ε, περιορίζει τα δικαιώματα των εμπλεκομένων στο δικαστήριο και εφόσον τα συμβαλόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν στην εφαρμογή του αποτελέσματος της διαμεσολάβησης δεν μπορεί να επιβληθεί. Η εμπιστευτικότητα δεν θεωρείται προβληματική από τα κράτη-μέλη. Ε, κλείνοντας να πω ότι ό,τι υπογραμμίζουν ότι υπάρχει διαφορά με τις χώρες τις οποίες η διαμεσολάβηση δεν ήταν παρούσα. Η οδηγία βοήθησε να υπάρξουν βήματα προόδου. Υπάρχουν ελάχιστες περιορισμένοι αριθμοί υποχρεώσεων για τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν προβλήματα ορισμών σοβαρά, υπάρχει μία κάποια εναρμόνιση σε σχέση με τις βασικές διαδικαστικές ειδικονομικές εγγυήσεις, υπάρχει ενθάρρυνση της διασφάλισης της ποιότητας και επίσης υπάρχει δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων. Η εμπειρία που έχει σωρευθεί μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε στο μέλλον εάν η οδηγία αυτή θα πρέπει να εμπνευστεί από το επίπεδο λεπτομέρειας της ADR. Αυτά. Merci beaucoup, Monsieur Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Τιμόσκι. Έχετε παρατηρήσεις οι υπόλοιποι συναδελφοί μου. Κύριε Χρυσόγονη. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συμμετέσχουν στην ακρόαση του Δεκεμβρίου σχετικά με την οδηγία για την διαμεσολάβηση. Τη θεώρησα πολύ καρποφόρα την ανταλλαγή απόψεων που διεξήχθη στην ακρόαση και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Χρυσόγανε. Ποιος επιθυμεί να παρέμβει εσείς κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβαση του κύριου Τιμόφσκι. Έχω μερικά γενικά σχόλια. Πρώτο, για την διαμεσολάβηση. Δεν είμαι βέβαια εχθρικός απέναντι στην διαμεσολάβηση. Είναι ένα τρόπος να λυθούν εξοδικαστικά ορισμένα, ορισμένες ε, διαφορές. Αλλά ούτε και μπορεί κανείς να την θεωρήσει πανάκια, διότι το δίκαιο εκδίδει κανόνες οι οποίοι κυρώνονται από τα δικαστήρια. Να μην προσπαθούμε να προωθήσουμε δε και καλά την διαμεσολάβηση, χάνοντας έτσι την βασική αυτή λειτουργία του δικαστηρίου. Γιατί το δικαστήριο έχει ως στόχο να αποκαταστήσει μια ισορροπία, μια ισότητα μεταξύ των μερών. Ενώ η διαμεσολάβηση δεν το πράττει αυτό. Η διαμεσολάβηση έχει πάντοτε την τάση να ευνοήσει τον ισχυρό απέναντι στον λιγότερο ισχυρό. Πολύ περισσότερο από ό,τι πράττει το δικαστήριο το οποίο αποκαθιστά την ισότητα. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη. Ο κύριος Τιμόφσκι εξέφρασε μια ενδιαφέρουσα άποψη. Είπε ότι υπάρχουν δύο γενναίες οδηγιών. Η πρώτη γενναία στην οποία κατατάσσει και την οδηγία διαμεσολάβησης, η οποία επιτρέπει μεγάλα περιθώρια ελευθερίας στην εφαρμογή από πλευρά των χωρών μελών, με τήρηση των παραδόσεων τους. Και μια δεύτερη γενναία, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε, η οποία δεύτερη γενεά επιβάλλει περισσότερες υποχρεώσεις στις ε, χώρες μέλη. είναι ε, πολύ σφιχτά τα όρια εκεί. Από την άποψη αυτή η οδηγία διαμεσολάβησης επιβάλλεται στις χώρες οι οποίες δεν ε, χρησιμοποιούσαν τη διαμεσολάβηση. Δεν είναι άσχημο αυτό, διότι τους δίνει μια πρόσθετη δυνατότητα επιλύσεως διαφορών, αλλά δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα από την επιτυχία αυτή ότι πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να αντικαταστήσουμε την ήπια αυτή οδηγία με μια οδηγία που θα είναι στην ουσία ένα κλουβί στο οποίο θα χωρέσουν μέσα οι ε, χώρε μέλη. Ευχαριστώ ε, αγαπητή κύριε κύριε Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ με τη σειρά μου τον κύριο Τιμόφσκι για την παρουσίαση που μου φάνηκε πολύ πλήρης ερώτηση για την Ιταλία η Ιταλία η οποία έχει καταστήσει υποχρεωτική την διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο και μόλις είπατε ότι έχουν αποφασίσει για λόγους διαδικαστικούς να το πράττουν αυτό. Μπορείτε να δώσετε κάπως περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν την ε, Ιταλία να θεσπίσει ως υποχρεωτική την ε, προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Σύντομα, πολύ σύντομα. Στη σελίδα 15 του εγγράφου μας λέμε ότι το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2012 απέριψε το διάταγμα όχι λόγω περιεχομένου αλλά λόγω τύπου και αυτό ανάγκασε την Ιταλική κυβέρνηση να επαναφέρει την υποχρέωση με ισχυρούς λόγους για να μπορέσει να αλαφρύνει από το μεγάλο βάρος το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Το έβαλαν όμως αυτό με μια ε, καταληκτική ρήτρα η οποία εξέπνευσε πέρσι. Δεν έχω ακούσει προτάσεις για να επαναληφθεί υποχρεωτικά η διαμεσολάβηση. Ακούω προτάσεις όμως, άλλωστε και στην ακρόαση, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να γίνεται μια πρώτη ακροματική διαδικασία υποχρεωτική για να αποφασίσουν τα μέρη αν επιθυμούν να προχωρήσουν στη διαμεσολάβηση. Γίνεται και κάποιο υπολογισμό κόστου με παραδείγματα από άλλε χώρε μέλη και με προβολή αυτού του αποτελέσματος και στι άλλες χώρε μέλη. Αλλά ίσως αυτό να μην στρέφεται οπωσδήποτε κατά ορισμένων παραδόσεων, αλλά νομίζω ότι μέσα από τις διάφορες πρακτικές που ακολουθούν οι χώρες μέλη μπορούν να επιλέξουν ορισμένες που μπορούν να ενταχθούν στα συστήματά τους. Η δεύτερη, επιτρέψτε μου να τη χαρακτήσω έτσι, γενεά των οδηγιών περιλαμβάνει διαδικαστικά στοιχεία πέραν της ε, οδηγίας διαμεσολαβήσεως. Καλή την πίστη με συμπερίληψη περισσότερων στοιχείων υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ο κύριος ε, Μαρίνιου Πίντου. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο μετά από τα όσα είπε ο συνάδελφος Λεμπρετών. Θέλω λοιπόν να πω ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης που έχει και υπάρχει σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να απομακρύνει τον κόσμο από τα δικαστήρια. Τα κράτη δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν να δεν έχει μάλλον παρά να οθήσει τους ανθρώπους, ε, τους διάδικους κάθε φορά να βρουν μία λύση ε, ειρηνική και πρέπει ωστόσο να τηρεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο της κάθε χώρας. Ε, η δικαιοσύνη επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τους πολίτες Όμως ε, πρέπει ε, μέσω διαδικασιών άλλων εποχών ε, γιατί θα ήθελα να πω ότι στι χώρες όπως η Πορτογαλία σε ένα δικαστηριό πρέπει να, στραφεί σε έναν δικαστή, σε κάνει εισαγγελέα Σχεδόν όπως ε, στην αρχαιότητα ένας δούλος απευθυνόταν ε, στον αφεντικό του. Ο πολίτης δηλαδή πιο εύκολα και πιο άνετα μπορεί να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της δημοκρατίας, με, τον έναν βασιλιά ή με μια βασίλισσα, από ότι μπορεί να μιλήσει με τον ε, εισαγγελέα ενός δικαστηρίου λόγω της μεγαλειώδους κατάστασης που επικρατεί. Και από την άλλη πλευρά, το δικαστικό σύστημα λειτουργεί πολύ άσχετα από τις αξίες και από τους, τους σύγχρονους καιρούς. Λειτουργεί περισσότερο σύμφωνα με τις δικές, τους, δικές του, του αξίες και τα σύμβολα και τη συμβολολογία άλλων εποχών. Ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται συχνά είναι ότι αν ένας πολίτης του καιρού της Γαλλικής Επανάστασης, για παράδειγμα, σήμερα πήγαινε σε μια πόλη στο Παρίσι ή στη Λισαβόνα, σίγουρα θα έμενε άναυδος με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία. Αν έμπαινε όμως το δικαστήριο στη Γαλλία ή στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, θα καθόταν και ήσυχα ήσυχα θα παρακολουθούσε μια κρεματική διαδικασία, γιατί από τότε στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η εσωτερική αρχιτεκτονική των δικαστήριων είναι η ίδια, τα ρούχα είναι τα ίδια, η, ε, η, αγορεύσεις είναι οι ίδιε, ε, υπάρχει μια δικαιοσύνη δηλαδή η οποία μένει εγκιστρωμένη σε σύμβολα άλλων εποχών και δεν έχει εξυγχρονιστεί. Και γι' αυτό και πολλέ φορέ το κράτο έχει δυσκολίε να διατηρήσει ή να συντηρήσει αυτή την δικαιοσύνη και προσπαθεί να φτιάξει εναλλακτικέ. Δηλαδή διπλασιάζει το κόστο και πολλέ φορέ και το χρόνο επίλυση των διαφορών. Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να είναι υποχρέωση του κράτου, πρέπει να είναι μια πρωτοβουλία των διαδίκων. Και εφόσον δεν μπορούν να βρουν λύση, τότε στρέφονται στο δικαστήριο. Μα γι' αυτό ε, στρέφονται στο δικαστήριο. Άρα λοιπόν το κράτος δεν χρειάζεται να τους υποχρεώνει να βρουν λύση. Ε, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φτάσει με δικαιοσύνη σε μια απόφαση η οποία σέβεται τις αρχές του κράτους, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης απέναντι στον νόμο, τις αξίες δηλαδή μια σύγχρονης δικαιοσύνης και όχι μιας πεπαλαιωμένης δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κομισιόν. Non Α, νόμιζα πως είχατε ζητήσει το λόγο. Δεν πειράζει, αφού δεν ε, θέλετε ή δεν μπορείτε. Περνάμε στην επόμενη φάση. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ περιορίστως και πάλι κύριε Τιμόφσκι και εσάς και την ομάδα σας για την ε, εισήγηση που μας κάνατε. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο σημείο 12 και το λόγο έχει ο συνάδελφος Χρυσόγονος. Uh. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πριν από 13 χρόνια το κανονισμό υπαριθμών 2006-2004 ε, σχετικά με τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, δημιουργώντας έναν μηχανισμό αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές προστασία του καταναλωτή. Υπ' αυτό το πλαίσιο οι αρχές ε, θα υποχρεούνται να ενεργούν εξ ονόματος ε, αλλήλων σε περιπτώσεις διασυνοριακών παραβάσεων. Ωστόσο, η, ανά, η ανάδυση παρακάμψεων διασυνοριακών ε, για το, στην νομοθεσία περί καταναλωτή ε, έφτασε στα όρια, της, ε, στα όρια του αυτόν τον κανονισμό. Έτσι η Κομισιόν ανταποκρίθηκε προτείνοντας αναθεώρηση του κανονισμού αυτού. Πρόταση που στόχο έχει να δώσει στα εθνικά όργανα προστασία του καταναλωτή περισσότερες αρμοδιότητες και να τους παροτρύνει να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους και μεταξύ άλλων ενώσεων όπως οι ενώσεις καταναλωτών. Επίσης θέλει να εξασφαλίσει την νομική βεβαιότητα στην ενιαία αγορά μέσω της συνεπούς επιβολής βασικών και εκτιμένων σχετικά με τον καταναλωτή που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα. Υπάρχουν ε, εθνικές ρυθμίσεις που δεν αρκούν για την επιβολή του εθνικού δικαίου περί καταναλωτή για να επιβληθεί διασυνοριακά το σχετικό δίκαιο. Άρα λοιπόν η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών είναι σημαντική ώστε να μην μπορούν οι έμποροι να ε, εκμεταλλεύονται παραθυράκια και κενά ε, σε κάθε κράτος μέλος. Ε, η πρόταση λοιπόν αυτή θα πρέπει καταρχήν να υποστηριχθεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα του καταναλωτή και να εξασφαλίζει ψηλό επίπεδο προστασίας του ιδίου. Πρέπει επίσης να ενεργεί προς την ασφάλεια των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή, να ενισχύει τα δικαιώματά του για την, ε, ε, στην ενημέρωση και την παιδεία, καθώς και να εξασφαλίζει τα συμφέροντά του. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πιθανή επιβολή αυτής της ε, νομοθεσίας, καθώς και στον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του καταναλωτή, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικό χώρο και στην προστασία των δεδομένων, πράγμα το οποίο είναι γεγραμμένο στο χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων Τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Επιπλέον, αυτό η πρόταση κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στην Οδηγία 9546 και στην, ε, στον κανονισμό 2016-679. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα υπό την εθνική τους νομοθεσία. Οι ενώσεις δε των καταναλωτών και οι ενώσεις, ε, εμπορικές ενώσεις ε, έχουν ασχοληθεί με τις ε, καταγγελίες των καταναλωτών, ιδιαίτερα στο ψηφιακό στην ψηφιακή αγορά. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα πλαίσιο για συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, προτροπές αυτών των ενώσεων ε, <coughs> που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6, εδάφιο 4 της πρότασης. Θα πρέπει λοιπόν να διαβουλεύονται και να αναζητώνται αυτές οι οργανώσεις και ενώσεις όταν αυτό χρειάζεται. Οι προτάσεις να λαμβάνονται απόψη στην ιεράρχηση των δράσεων επιβολής. Επιπλέον σε περίπτωση που μια παράβαση ε, επαναλαμβάνεται και χρειάζονται νέα με, περαιτέρω μέτρα, εγώ θα σύστηνα η αρμόδια αρχή να ενημερώνει την Κομισιόν και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών χωρίς καθυστέρηση έτσι ώστε να μπορεί άμεσα να προβεί σε ενέργειες. Επιπλέον συστήνεται να διευρυνθούν οι απαιτήσει ε, για δεδομένες ε, παραβάσεις ε, με ανθρώπινη διάσταση. Εκεί όπου υπάρχει υποψία, όπου κάποια διαδεδομένη παράβαση ε, πρόκειται να βλάψει ή θεωρείται ότι θα βλάψει καταναλωτέ στα μισά κράτη-μέλη, που μαζί αποτελούν τουλάχιστον το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ένωσης, η Κομισιόν θα ξεκινήσει κοινέ ενέργειε ώστε να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές των καταναλωτών να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών στην Ένωση εκεί όπου η προτινόμενη δράση δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα κράτος μέλος μόνο του και έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως ε, θα επιβληθούν σωστά οι νομοθεσίες περί καταναλωτών, περί προστασίας του καταναλωτή. Επιπλέον, θα υποβάλλεται έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, το αργότερο μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύω της εφαρμογής αντί για τα 7 χρόνια που ε, αρχικά πρότεινε η Κομισιόν στην πρότασή της. Δεδομένων των διαφορετικών προσεγγίσεων ε, επιβολής και ε, σε κρατημέλη, πράγμα το οποίο καταλήγει σε διαφορετικές απαντήσεις, σε παρόμοιες ή και ίδιες παραβάσεις, ίσως και καμία απολύτως απάντηση, Πολλές φορές αυτό οδηγεί στην απαξίωση της ενιαίας αγοράς στα μάτια των καταναλωτών. Κεντρικός ρόλος της Κομισιόν όσον αφορά την οδιοργάνωση της συνεργασίας ανάμεσα στις ε, εθνικές αρχές και την επιβολή των, ε, της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή θα πρέπει να προωθηθεί. Ο ρόλος των ε, και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή θα πρέπει να τονιστεί ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο ρόλο της Κομισιόν και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών υπέρ πάντοτε της προστασίας του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυσόγονε. κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την θαυμάσια γνωμοδότηση. Συμφωνούμε με τον στόχο της προτάσεως γνωρίζουμε όλες και όλοι ότι έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την επιβολή των διατάξεων του νόμου είναι διαφορετική. Και ιδίω αυτό αποτελεί πρόβλημα σε διαμεθοριακές υποθέσεις. Για παράδειγμα, παραβιάσεις διατάξεων προστασίας του καταναλωτού στον, στην ψηφιακή αγορά. Για να επιτευθεί πρόοδος στην υπόθεση αυτή, θα πρέπει να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, των φορέων δηλαδή προστασία των καταναλωτών μεταξύ των διαφόρων χωρών. Εμεί εγκρίνουμε και να αναλάβει ένα ισχυρότερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη των ευριών παραβιάσεων που ε, πιάνουν πολλέ χώρε μέλη τη Ένωση και ταυτόχρονα νομίζουμε ότι αυτή η κοινή διαδικασία δεν καθορίζεται με επαρκή λεπτομέρεια στην πρόταση. Πολλές λεπτομέρειες ε, ανατίθενται να ρυθμιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εφαρμοστικές πράξεις και νομίζουμε ότι ιδίω σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη γνωμοδότηση του εισηγητού είναι σημαντικό και εκεί να εμπλουτιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες δηλαδή σχετικά με την αναστολή λειτουργίας ιστοσελιδών ή ιστοχώρων συνολικότερα, εκεί νομίζουμε ότι αυτό έχει τεράστια επίπτωση στην ελευθερία του λόγου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εγγύσεις πρώτα πριν να ανασταλεί η λειτουργία ενός ιστοχώρου και θα πρέπει να υπάρχει και δικαστική απόφαση. Εξάλλου θεωρούμε ότι η ενεργός συμμετοχή Τη κοινωνία των πολιτών, των ε, φορέων προστασία των καταναλωτών, που συχνά δεν είναι κρατικέ αρχέ, θα πρέπει και αυτή να ενισχυθεί για να μπορέσει να αποδώσει η στρατηγική προστασία των καταναλωτών εν τέλει. Σημαντικό είναι επίση όταν θα κριθεί ποιο φορέας θα είναι αρμόδιο για να ηγηθεί, για να λάβει δηλαδή τον πρωταρχικό ρόλο, διότι βεβαίω οι πόροι που απολαμβάνουν οι διάφοροι φορείς από χώρα σε χώρα είναι πολύ διαφορετικοί χρειάζεται και εκεί συνεργασία. Και οι χώρες μέλη θα πρέπει να φέρουν τους φορείς προστασίας καταναλωτών σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να έχουν επομένως επαρκείς πόρους. Εν τέλει, σε ό,τι αφορά το παράρτημα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να περιλάβουμε ήδη κάποιες από τις νομοθεσίες προστασίας καταναλωτών που ήδη λειτουργούν καλά και που μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα, όπως ο κανονισμός για τη δυνατότητα μεταφοράς. Μπορεί να μπει στο παράρτημα. Θα αρκεστώ σε αυτά. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία που έχει ήδη επιτελέσει και θα συνεργαστώ ευχαρίστω μαζί του για τη συνέχεια. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα επανέλθω στον συνάδελφό μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον εισηγητή για την πολύ θετική έκθεση. Καθώς επίσης και την κυρία Ρέντα για την παρέμβασή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι έχει καταθέσει πρόταση για την ενίσχυση των υφισταμένων μηχανισμών του υφισταμένου μηχανισμού, που ωστόσο έχει ορισμένες αδυναμίες. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ε, ε, ευρείας εφαρμογής παραβιάσεων, να το πω έτσι, και της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών όλων των χώρων μελών της Ένωσης. Εμείς προτείνουμε ένα μηχανισμό όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τον ρόλο να καθορίζει τους όρους για την εκκίνηση μιας συντονισμένη δράσεως όταν αυτή θα αφορά μέγα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό έχουμε βάλει κατόφλια και τα κατόφλια αυτά είναι το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 75% των ευρωπαϊκών χωρών, των μελών, χωρών μελών δηλαδή τη Ένωσης. Γιατί βάζουμε τόσο υψηλά το κατόφλι, διότι θεωρούμε ότι μόνο σε τέτοιε περιπτώσει είναι πράγματι αναλογική η προσέγγιση αυτή και σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Το να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ρόλο αυτό. Να ζητήσει από τις χώρες μέλη δηλαδή να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις δράσεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε υποθέσεις που είναι κάτω από το κατόφλι αυτό δεν θα παίξει τον συντονιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα εξαρτηθεί από τις υποθέσεις και θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες των χωρών μελών να οργανωθούν μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει βέβαια με θετική ε, πρόθεση όλες τις ε, συντονισμένες δράσεις. Θα πρέπει όμως να ε, συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ιδίως στα θέματα εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στην ενιαία αγορά. Σε ό,τι αφορά την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, το δικαίωμα των καταναλωτού, τη προστασία του καταναλωτού δηλαδή, είναι και αυτό ένα θεμελιωδή δικαίωμα. Το ερώτημα είναι, το ζήτημα μάλλον είναι να βρεθεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στι διάφορε αξίε των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το δικαίωμα του ελευθέρω επιχειρήν, την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτού. Και νομίζουμε ότι στα πλαίσια τη ενιαία ψηφιακή αγορά είναι σημαντικό οι παραβιάσει του δικαίου προστασία του καταναλωτού να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο. Γιατί? Διότι μπορεί να υπάρχει ένας ε, έμπορος, απαταιώνας έμπορος ο οποίος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και βγάζει πολλά λεφτά στην πλάτη των καταναλωτών προτείνοντας υπηρεσίες τις οποίες δεν παρέχει ποτέ ή προσελκύοντας τους καταναλωτές να εγγραφούν συνδρομητές σε πράγματα τα οποία δεν ήθελαν. Δεν υπάρχει κατάστημα, του εμπόρου αυτού, ε, κινείται όπου θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον λόγο αυτό προτείνουμε οι χώρες μέλη να έχουν την εξουσία να εμποδίζουν την πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή στο συγκεκριμένο ψηφιακό περιεχόμενο, κυρίως για να μπορέσει να κοπεί ο δρόμος σε τέτοιες απάτες. Όσον αφορά την διαδικασία που εφαρμόζεται στις χώρες μέλη, αυτή πρέπει να γίνει σεβαστή. Ο κανονισμός CPC βασίζεται στον σεβασμό των διαφόρων διαδικασιών που χρησιμοποιούνται τώρα στις χώρες μέλη και οι διαδικασίες αυτές που ήδη ευθυγραμμίζονται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν πολλές εγγύησεις. Όμως, για να γίνει σαφέστερο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει να εισαχθούν να εγκριθούν ε, άλλα στοιχεία του κειμένου για να φανεί καθαρά, προτείνει μάλλον να προεδρευτούν και άλλα στοιχεία του κειμένου για να φανεί καθαρά ότι ε, γίνονται σεβαστά τα, δικα, τα διαδικαστικά δικαιώματα, βεβαίω οι συνταγματικέ διατάξει και τα ε, δικαιώματα των εμπόρων. Όσον αφορά το ενδεχόμενο να περιληφθεί πρόσθετο κείμενο στο παράρτημα, εάν αυτό θα αφορά κείμενα τα οποία συζητούνται τώρα, αυτά πρέπει να συζητηθούν μέσα στο πλαίσιο του παρόντος θέματος. Αν εξετάσετε για παράδειγμα τον κανονισμό για το γεωγραφικό αποκλεισμό που θα εξετάσουμε αμέσως μετά, περιλαμβάνει διάταξη σχετική με την επιβολή κανόνων για προβλήματα που ε, συμβαίνουν μεταξύ επιχειρήσεων και, και ε, πελατών και καταναλωτών. Αν δείτε άλλους, άλλα κείμενα θα δείτε ότι υπάρχει από παρόμοιοι κανόνες, αλλά για business του consumer πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο, διότι ο κανονισμός CPC, στην πρώτη περίπτωση γίνεται παραπομπή στον CPC, κανονισμό αυτό δεν μπορεί να γίνεται παραπομπή σε άλλη νομοθεσία η οποία δεν υφίσταται ακόμη. Είναι ζήτημα δηλαδή νομικοτεχνικό. Έτσι πρέπει να γίνει. Βεβαίω, ευχαρίστω θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια ευρωβουλευτών οι οποίοι θα ήθελαν να υποβάλλουν τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος όχι, με συγχωρείτε επανέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσθέσω κάτι ακόμη για τις οργανώσεις καταναλωτών και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση των οργανισμών αυτών. Βεβαίω εμείς είμαστε υπέρ, υποστηρίζουμε οργανώσεις προστασίας καταναλωτών μέσω του προγράμματός μας, Consumer Program, και είναι σημαντικό για μας οι διατάξεις που έχουν σχέση με τη δυνατότητα των φορέων προστασίας καταναλωτών ε, να ε, βγάζουν μηνύματα ε, για τους καταναλωτές κλπ. Περιλαμβάνεται στις προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Γουόγκα. Να μην υπάρξει διάκριση σε βάρος των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τους τρόπους πληρωμής. νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβετε, διότι υπήρξε μια ε, σύντομη διακοπή του μικροφόνου σας. Επαναλαμβάνει ο κ. Γκόγκα. Ήθελα να απευθυνόμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει διάκριση σε βάρος ε, πελατών μόνο και μόνο λόγω του τρόπου πληρωμής των οποίων έχουν επιλέξει. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Υποθέτω ότι είναι ένα σχόλιο το οποίο απευθύνεται περισσότερο στον εισηγητή, δεν είναι δηλαδή ερώτηση προ την Κομισιόν. Δεν αναμένεται ε, απάντηση, έτσι είναι. Όχι, όχι, δεν αναμένω απάντηση, ε, απάντησε ο κ. Γκόγκ. Απλώ ε, επισημαίνω μια παρατήρηση. Ο κ. Λεμπρετών. Δεν είχα την πρόθεση να λάβω το λόγο για το θέμα αυτό, αλλά θα κάνω σύντομο σχόλιο. Πρώτα να πω ότι η κυρία Ρέντα καλά λέει ότι εάν πρόκειται να ανασταλεί ε, η χρήση κάποιων ιστοσελίδων πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγγύησεις διότι πρόκειται για την παρέμβαση στην ελευθερία του λόγου και νομίζω ότι χρειάζεται όντως παρέμβαση δικαστού. Δεύτερον, ομολογώ ότι κατεπλάγει από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή όλα πάνε καλά, είπε κάποια τεχνικά πράγματα τα οποία σέβομαι εκτός πια και αν υπάρχει πρόβλημα μεταφράσεως, ε, διότι προτείνει την βοήθειά της για να συντάξουμε τροπολογίες. Ευτυχώς που καθόμουν, διότι θα είχα πέσει κάτω. Η δουλειά του Ευρωβουλευτού είναι να συντάσει τις τροπολογίες του ο ίδιος μόνος του. Εάν για να τροπολογήσει ένα κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να προσφύγει στην βοήθεια της Επιτροπής, ε, τότε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε τότε να πάμε σπίτια μας και να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πάντα μόνη της. Να ψηφίσει κιόλας. Ειλικρινώς, δεν νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τέτοιο δρόμο. Θεωρώ ότι ήταν μια πρόταση καλής προθέσεως. Δεν υπάρχει πρόταση εκ μέρους σας. Ε, Λαμβάνει το σχόλιο όσο έχει. Ευχαριστώ. Εσείς τώρα κύριε Σιγητά θέλετε να ολοκληρώσετε. Uh, I would just like to thank uh, everybody. Εγώ θέλω μόνο να ευχαριστήσω όλες και όλους που συμμετέσχουν στην γόνιμη αυτή συζήτηση και θα προχωρήσουμε και θα σας ειδοποιήσω. Merci beaucoup. Je rappelle... Σας ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 13. Η κυρία Γκέριγκερ Ντεόρντεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας αναφερθώ στο, στο γεωγραφικό αποκλεισμό στο geo-blocking και σε άλλες μορφές ε, διάκρισης που δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τον τόπο κατοικίας, τον τόπο εγκατάστασης ε, ή και στον τόπο ακριβώς διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο κανονισμός για το geo-blocking ε, έχει στόχους υπέρ του καταναλωτή αλλά και υπέρ των επιχειρήσεων λέγει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες και επιλογές. Από την άλλη βοηθά τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις δραστηριότητες τους εφαρμόζοντας στους ξένους πελάτες ε, την υποχρέωση της μη επιπλέον δημιουργίας διακρίσεων. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να ελέγξουμε κάπως καλύτερα για να πετύχει τους στόχους του ο κανονισμός. Τώρα για τους καταναλωτές. Εδώ θα έλεγα είναι πολύ σημαντικός ο όρος geo-blocking, σημαίνει το απαγόρευση πρόσβασης σε ε, πολιτιστικά προϊόντα, αθλητικά γεγονότα ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο γεωγραφικός αποκλισμός, ε, είναι κάτι το οποίο δεν ορίζεται καταρχάς στους όρους διανομής ενός προϊόντος. Καλύπτεται εδώ ο, με ηλεκτρονικό τρόπο, θα έλεγα, ο, με ηλεκτρονικό τρόπο διαδικασία διάδοσης του προϊόντος και αναπαραγωγής του προϊόντος. Σαν στόχος κάτι τέτοιο ακούγεται λίγο περίεργο και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω την διεύρυνση του άρθρου 4 της πρότασης έτσι ώστε να σε περιλάβουμε και τα ε, e-books και τα video games και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. καλύπτεται από τον κανονισμό λοιπόν εφόσον ο διανομέας έχει τα δικαιώματα διάδοσης στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια του έργου. Αυτό λέγει και το άρθρο 9. Ε, το geo-blocking έχει σαν στόχο και την διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας έχει σαν στόχο την προστασία της δημιουργικής, αν θέλετε, πλευράς της δραστηριότητας. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τους καλλιτέχνες και δημιουργούς ή να διαφοροποιήσω την κατηγορία τους σε σχέση με άλλους παραγωγούς προϊόντων. Αλλά η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σαν παράδειγμα πολλοί Πολωνοί πολίτες, Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί κατοικούν σε διαφορετικές χώρες. Και γι' αυτό θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση ε, ε, σε έργα της χώρας και της γλώσσας από την οποία προέρχονται. Έχουμε ξεκινήσει και εμείς οι ίδιοι ιστοσελίδες στις χώρες μας. Όταν θέλουμε να διαβάσουμε κάτι στη χώρα μας, πατάμε την ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν είμαστε στη Μάλτα ή στο Βέλγιο δεν μπορούμε να δούμε το συγκεκριμένο προϊόν ε, λόγω των προβλημάτων του copyright. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα βήμα φιλόδοξο να έρθουμε πιο κοντά στους ε, ε, συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν το θέμα του geo-blocking. Τώρα, αυτά για τους καταναλωτές. Να δούμε τώρα για τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι το ότι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις συμβάσεις. Θα είναι ο νόμος της χώρας στην οποία ε, έχει την έδρα της η επιχείρηση ή ο νόμος της χώρας, ο οποίος, ε, της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο καταναλωτής. Για τις καταναλωτικές συμβάσεις ε, ο νόμος της χώρας όπου κατοικεί ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Αυτό προβλέπεται από την άλλη να έχουμε υπόψη μας ότι ε, ο κανονισμός για τον τερματισμό του γεωγραφικού αποκλεισμού περιορίζει την ελευθερία των δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών επιβάλλοντας την μη διάκριση εις βάρος των ξένων καταναλωτών. Είναι λοιπόν και πρέπει να είναι η επιχείρηση ελεύθερη να ε, συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις με οποιονδήποτε και οπουδήποτε το επιθυμεί. Συνεπώς λοιπόν ο κανονισμός θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στις επιχειρήσεις και να προστατεύσει καλύτερα α, ε, τις δραστηριότητές τους. Ε, νομίζω λοιπόν ότι εμείς δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν α, συνεργαστεί στο επίπεδο το οποίο θα επιθυμούσαν και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο το νομικό καθεστώς της χώρας τους αλλά και των υπολείπων 27 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν μια χώρα σαν παράδειγμα αποκλειστικά έχει στο νου της καταναλωτές μία συγκεκριμένης χώρας, τα λεγόμενα targeted sales, στοχευμένες πωλήσει, τότε ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτόν για τον καθορισμό του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο ε, ε, γίνεται η δραστηριότητα αυτή. Όταν η πλειοψηφία των πελατών προέρχεται από μία χώρα, τότε η χώρα των καταναλωτών θα είναι αυτή η οποία θα παρέχει το νομικό πλαίσιο. μέσω της ε, ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας ε, επιχειρηματικής ο καταναλωτής συμφωνεί στα πλαίσια της υπογραφής της συμφωνίας ε, με το νομικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει. Πρέπει λοιπόν η νομική ρύθμιση να προστατεύει τον καταναλωτή και όταν κάποιος αγοράζει στο Βέλγιο κάτι από την Πορτογαλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πρέπει να προστατεύεται ως προς αυτό. Εγώ δεν θα ήθελα οι επιχειρήσεις μας να γνωρίζουν, να κατέχουν 27 διαφορετικά νομικά συστήματα. Αλλά θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ε, και να μην ε, ε, προχωρούν σε συμφωνίες αγορών κτλ οι οποίες για αυτούς παρουσιάζουν δείγματα ανασφάλειας σε σχέση με το νομικό τους πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν βάση και στους επιχειρηματίες, κυρίως όμως τους καταναλωτές. Πρέπει να έχουν ευρύτατη πρόσβαση στα, στην πολιτιστική δημιουργία, όχι άμεσα αλλά σταδιακά. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τις επιλογές αυτές, αλλά όχι όμως αυτό να επιβαρύνει γραφειοκρατικά τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα ήθελα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουδήποτε άλλου συναδέλφου. Η κυρία Ρέντα, ή μάλλον πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μου το επιτρέπει η κυρία Ρέντα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ο εκπρόσωπος. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά. Η πρόταση προσπαθεί να εξισορροπήσει τα θεμητά συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις αδικαιολόγητες μορφές διακρίσεων. έτσι ώστε να μην υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να μην εξυπηρετούν καταναλωτές οι οποίοι με τη σειρά τους θα απογοητευόντουσαν από αυτήν την έλλειψη δυνατότητας. Αναφερόμαστε κυρίως στο δημιουργικό περιεχόμενο ε, πολιτιστικών έργων, οπτικοακουστικής φύσεως. Ήδη είχαμε πει ότι εμείς θέλουμε μετά από τις ρυθμίσεις που είχαμε περάσει να υπάρξει μια αναθεώρηση μετά από ένα χρονικό διάστημα. Και εσείς είπατε ότι θα θέλαμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι επιπτώσεις είχε η ε, νομοθετική ρύθμιση την οποία είχαμε περάσει και τι ακριβώς έχουν να κερδίσουν οι καταναλωτές αυτοί. Γιατί ιδιαίτερα για τον μη οπτικοακουστικό τομέα είχαμε πολύ λίγα στοιχεία για τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής του geo-blocking. Αυτό δεν είναι μια δήλωση υπέρ κατά του geo-blocking, δεν είναι ιδεολογικά φορτισμένη θέση. Θα θέλαμε να δούμε ακριβώς πώς συμπεριφέρονται οι αγορές μουσικών προϊόντων. Τα θέματα αυτά δεν συνδέονται μόνο με το θέμα της προστασίας του copyright. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις, οι μουσικές έχουν τα δικαιώματα για το σύνολο του καταλόγου τους, για το σύνολο των χωρών. Είναι περισσότερο θέματα επιχειρηματικά και θα πρέπει να δούμε ακριβώς αν τους ζητήσουμε να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, τι θα αλλάξει για τους καταναλωτές ιδιαίτερα στον τομέα της τιμολόγησης των προϊόντων. Η έκκλησή μας λοιπόν είναι να υπάρξει μια συζήτηση αυτών των θεμάτων. Προς το παρόν ε, συλλέγουμε στοιχεία για να τροφοδοτήσουμε τον τριμερή διάλογο στον οποίο θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Ε, το θέμα αυτό έχει συζητηθεί και στο Συμβούλιο. Βασική θέση μας είναι ότι δεν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε τα συστήματα προστασίας του καταναλωτή στις διάφορες χώρες. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι εμείς ζητάμε από τους εμπόρους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα αιτήματα παροχής υπηρεσιών και σε άλλες χώρες όλο και περισσότερο. Και θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι το να είναι συμβατή λειτουργία τους με τον κανονισμό αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να στρέψουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες υποχρεωτικά. Αλλά θέλουμε να διευκρινίσουμε ε, ότι όταν ένας έμπορος ασκεί δραστηριότητες και σε άλλες χώρες θα πρέπει να εφαρμόζεται η σωστή νομική βάση. Θέλουμε δηλαδή να διευκρινίσουμε την κατάσταση και μάλιστα το Συμβούλιο έκανε περαιτέρω βήματα προόδου χωρίς να αλλάξει τις ε, υποβόσκουσες αρχές, αν θέλετε, αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, προσπάθησε να ορίσει το ποιες είναι οι δραστηριότητες δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την νομική ρύθμιση και φυσικά ζητήσαμε και με το Κοινοβούλιο για το πώς ακριβώς θα γίνουν οι διακρίσεις αυτές και περιμένω και εγώ με τη σειρά μου τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του, ε, της, ε, ε, το εξαιρετικό της σχέδιο γνωμοδότησης. Ήδη βλέπουμε στο σχέδιο έκθεσης αρκετή σύγκληση με τις συζητήσεις που γίνονται και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. το θέμα του γεωπεριορισμού είναι σημαντικό. Είναι κάτι που το ζητά ο κόσμος. Ζητά περισσότερη Ευρώπη και περισσότερες λύσεις και δεν καταλαβαίνουν πώ στην ενιαία αγορά μπορεί κανείς να ορθώσει τεχνητά σύνορα στο ίντερνετ. Γι' αυτό και καλωσορίζω τη φιλοδοξία της εισηγήτρια να επεκτεθεί το πεδίο εφαρμογή. Είναι ωστόσο εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν ο κόσμο ακούει για περιορισμό περισσότερο σκέφτεται βίντεο, τα βίντεο. Πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα του οπτικοακουστικού περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα αν κάποιοι συνάδελφοι αρχίζουν να ανησυχούν όταν τα ακούν όλα αυτά, είναι σημαντικό πιστεύω να γνωρίζουμε ότι αυτό που προτείνει η συγγήτρια είναι να συμπεριληφθούν τα το περιεχόμενο ε, με copyright εάν υπάρχει, αν ο πολιτής έχει άδεια. Το θέμα του Copyright θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την νομοθεσία περί copyright. Εδώ Μιλάμε για γεωπεριορισμούς που επιβάλλονται για λόγους εκτός copyright, όταν υπάρχουν, όταν έχουν χορηγηθεί άδειε. Η Κομισιόν θα πρέπει να δει επίσης την εργασία που έχει ήδη γίνει ε, σε αυτό το θέμα. Ας πούμε για την ε, δυνατότητα ε, φορητότητας στη σχετική οδηγία έχουμε βρει ότι υπάρχει ήδη εκτεταμένη παγκόσμια διοδότηση και στον ε, τομέα του αθλητισμού όταν δεν έχει να κάνει με τα premium όπου οι ε, εδαφικές ε, άδειες είναι πολύ συγκεκριμένες γιατί λοιπόν να μην το επιτρέπουμε στους πολιτές εφόσον το copyright δεν είναι εμπόδιο. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, επέκταση του πεδίου εφαρμογή και καλό την Κομισιόν να δει και τι έχει γίνει στις υπόλοιπες σχετικές όμως, ε, στους υπόλοιπους σχετικούς τομείς νομοθεσίας. Επίσης είναι καλό το ότι η συγκήτρια αφήνει επαφές σε τις αρχές τη... στις αρχές της Κομισιόν για τις, ε, ε, για τις ε, επιγραμμικές προσφορές, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν εταιρείε που πολλούν διασυνοριακά. Και δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα παραθυράκι όπου να μπορούν να πούνε εμείς δεν ακολουθούμε πλέον τον νομοθεσία καταναλωτή των άλλων χωρών επειδή υπάρχει ο κανονισμός για, για τους γεωπεριορισμούς. Ίσως λοιπόν θα πρέπει στα recitals να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς γίνεται σε περιπτώσεις όπου ο πολιτής δεν θεωρείται ότι στοχεύει άλλες χώρες. Ίσως αυτό θα είναι μια βιώσιμη προσέγγιση και ίσως θα είναι πιο ωφελική προς τον καταναλωτή από αυτό που βλέπουμε στο σχέδιο εκθέσης της ΙΜΚΟ για την ώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι εργαζόμαστε επί τη βάση ενός πολύ καλού κειμένου και ότι θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος σύντομα. Είναι κάτι όπου οι καταναλωτές θα ωφεληθούν, θα έχουν προσθέμενη αξιά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαντεύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ την κυρία Γκέριγκερ για την ε, πολύ ισορροπημένη γνωμοδότηση. Πολλοί έμποροι ε, κάποιων χωρών μελών εξακολουθούν να μπλοκάρουν ή να παρεμποδίζουν την πρόσβαση ε, στα site τους ε, για πελάτες άλλων χωρών μελών. Τεχνητός περιορισμός της αγοράς και περιορισμός της επιλογής των καταναλωτών. Η πρόθεση των καταναλωτών προς ενδιάμεσους οδηγεί σε παραπάνω κόστος. Κάποιες φορές υπάρχουν κάποιοι όροι που να δικαιολογούν διαφοροποιημένη μεταχείριση, όμως συχνά οι έμποροι αρνούνται την πρόσβαση στο site τους σε αλλοδαπούς πελάτες για απλά εμπορικούς λόγους και τη απουσία υγιούς ανταγωνισμού. Ορισμένοι έμποροι χρεώνουν υπερβολικά τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να συντάξουμε πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία που θα επιτρέπει διαφοροποιημένη μεταχείριση ώστε να, υπάρξει, να επικρατήσει μάλλον μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για όλους και ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την εφαρμογή κανόνων μη διάκρισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξεχνάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην τις επιφαρύνουμε με τεράστιο διοικητικό φόρτο ε, στη θέματα των διασυνοριακών συναλλαγών. Η οικονομία και ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα του γεωπεριορισμού οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στην καλύτερη τιμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκούγκα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Αποτελεί μια ε, καλή βάση για περαιτέρω συζητήσει. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε νομική σαφήνεια και να αποφύγουμε περιστάσεις όπου θα επικρατούν αμφιβολίες για το πώ θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες. Η διατύπωση για το εφαρμοστέο δίκαιο ε, είναι, επιδέχεται βελτίωση. Και για την πιθανή επέκταση πιστεύω πως η Κομισιόν δεν στάθη αρκετά φιλόδοξη όταν πρότεινε να επιθυγραμμιστεί το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση προ την οδηγία περί υπηρεσιών, γιατί αποκλείονται κάποιε δραστηριότητε όπω οι υπηρεσίε μεταφορά και οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Τούτου λεχθέντο, θα πρέπει να πω ότι κάθε επέκταση πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση αποδείξεων, αποδεικτικών στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να ξανατονίσουμε την μη διάκριση αντίον των, πελατών με βάση το τρόπο πληρωμής. Ας Δηλαδή να μην γίνονται διακρίσεις ε, στους ε, πελάτες ανάλογα με το ποιο τρόπο χρησιμοποιούν για την πληρωμή. Στο άρθρο 5 Τώρα ε, δεν έχουν γίνει τροπολογίε. Εγώ θα προτείνω σχετικέ και προσβλέπω συνεργασία με του συναδέλφου τη Επιτροπή ώστε να βρούμε τι καλύτερε λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την παρέμβασή σα, Ο κύριος Λεμπρετό. Ε, Κάποιε γενικές παρατηρήσεις έχω να κάνω. Κατανοώ τα όσα υπόθηκαν για να δικαιολογηθεί ο, ο σε ορισμένου τομεί. Εγώ ε, θα είμαι ο συνήγορος του διαβόλου για να πω ότι εφόσον υπάρχουν γεωπεριορισμοί. Αυτό δεν ε, είναι μόνο για προς χάρη διοικητικού φόρτου, ε, ε, είπαν κάποιοι ότι οι καταναλωτές ενοχλούνται διότι έχουν να κάνουν με 27 διαφορετικά νομικά συστήματα και οι επιχειρήσεις επίσης δυσκολεύονται, αλλά πρέπει αυτό να μας κάνει καχύποπτους, γιατί ε, αν το πάμε έτσι θα καταργηθεί τελείως το εθνικό δίκαιο. Είναι λογικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλού και όχι μόνο στο γεωπεριορισμό, γιατί υπάρχει, γιατί οι καταναλωτές δεν είναι μόνο οι πολίτες δεν είναι μόνο καταναλωτές. Έχουν τις εθνικές τους παραδόσεις, θέλουν η εθνική τους οικονομία να προστατεύεται σε ορισμένους τομείς. Επίσης, ε, είναι μια θεμητή ανησυχία που πρέπει να γίνει σεβαστή και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σας προειδοποιήσω εναντίον μιας παράλογης επέκτασης της Κομισιόν. Η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει προσεκτικά, έχει δίκιο και εμείς δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε γιατί ακόμα μια φορά θα είμαστε απομακρυσμένοι από τις επιθυμίες των λαών μας. Σας ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από τους συναδέλφους, θέλω και εγώ να σας δώσω τη γνώμη μου ως μέλος της Επιτροπής και όχι ως πρόεδρος. Προεδρεύων μάλλον αυτή τη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ καταρχά, κυρία Σιγήτρια, για την εργασία σα. Εσεί και η ίδια ε, κάνατε πολύ ε, καλή δουλειά. Να πω ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο εν τη σοφία τους έχουν δίκιο να μην λαμβάνουν υπόψη σε αυτή την πρόταση κανονισμού ε, τα περιεχόμενα που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα γιατί, θα, ε, γιατί φαίνεται προφανές ότι το να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση θα σήμαινε να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, από, το οποίο δεν, από την οποία συζήτηση πρόκειται να βγούμε χωρίς σημαντικές ζημιές. Οπότε, γι' αυτό και σας συγχαίρω για αυτή τη μετρημένη προσέγγιση. Ε, θα έχουμε το χρόνο να το εξετάσουμε και πιστεύω πως είναι ο καλύτερος τρόπος να νομοθετούμε και να ασκούμε τον έλεγχο όσο γίνεται πιο νυφάλια ως κοινοβούλιο. Να πω ακόμα κάτι ουσιαστικό ε, που ε, εγώ υποστηρίζω ως ιδέα, ότι δεν πρέπει να αμφισβητηθούν οι κανόνες σε θέματα προστασίας ε, πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Αλλά να πω αντίθετα ότι δεν μπορώ να μείνω ικανοποιημένο από αυτή την προσέγγιση που συνίσταται στο να αναβάλουμε σε μια περαιτέρω μεταγενέστερη μάλλον αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικώς για τα έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, τον τρόπο διανομής τους. Αν αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνει, θα ήθελα να γίνει εις βάθος, όπως ε, είπατε κι εσείς ε, ότι πρέπει να γίνει, και να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των έργων που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτά είναι πηγή κάθε δημιουργίας και είναι και το συμφέρον αυτών που έχουν πλατφόρμες να έχουν διαφοροποιημένη προσφορά σε αυτό το τόσο πλούσιο ε, περιβάλλον προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πνευματικά δικαιώματα λοιπόν στους διάφορους ε, ε, Τομεί πνευματική δημιουργίας που επιτρέπει την ε, χρηματοδότηση και συντηρίζω τη δίκαια αμοιβή των ε, δημιουργών γιατί αυτό είναι η βάση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και μπορεί να εξασφαλίσει ε, εσαΐ την πολιτιστική δημιουργία. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτές οι υπηρεσίες να προστατευτούν και αυτό θα το προσπαθήσουμε. Η αρχή τώρα της εδαφικότητας επιτρέπει να αποφύγουμε τη συγκέντρωση κυρίαρχων φορέων στην αγορά εις βάρος των ελλακτικών προσφορών και ε, των όσων δεν έχουν τα ίδια οικονομικά μέσα και κυρίως εις βάρος των ανεξαρτήτων που είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την προσφορά της διαφορετικότητας γιατί όσο πιο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις, οι όμιλοι τόσο μειώνεται η διαφοροποίηση και η διαφορετικότητα. Το βλέπουμε σε όλους τους τομείς και επίσης πολύ στον τομέα του πολιτισμού. Να θυμίσω ότι ο κανονισμός για τη φορητότητα, για τον οποίο ήμουν εισηγητής και όπου η Νομική Επιτροπή ναι, έκρινε την έκθεσή μου ομόφωνα στα τέλη του περασμένου έτους, ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα του γεωπεριορισμού που δεν, που, που δεν δικαιολογούνται ε, για θέματα περιεχομένου στα κράτη-μέλη. Τώρα, Όσον αφορά την καταπολέμηση των γεωγραφικών διακρίσεων, αυτό είναι μια πολύ καλή ε, ιδέα. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και επίσης για ό,τι μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία τους χωρίς να, επηρεάζεται, ε, να επηρεάζονται οι βασικές αρχές ε, να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, αλλά σοβαρά με πραγματική βούληση ενοποίησης όσων μπορούν να ενοποιηθούν. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρξουν καταχρήσεις και να αντιδρούμε εφόσον δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος που να αιτιολογεί τη ε, γεωγραφική διάκριση. Και από αυτή την άποψη στηρίζω τη δική σας προσέγγιση. Ωστόσο είμαι πεπισμένος ότι η καταπολέμηση των γεωγραφικών διακρίσεων, των αδικαιολόγητων, ε, σημαίνει τη βελτίωση της δυνατότητας του καταναλωτή να εντοπίζει αλλά και να υπεραμείνεται το αυτού του εναντίον αυτών των διακρίσεων. Για να το καταφέρουμε αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαφάνειας απέναντι στον καταναλωτή αλλά και να ενισχύσουμε την ενημέρωσή του. Θεωρώ επίσης πως πρέπει να ε, παγρυπνούμε εναντίον κάθε απόπειρας κατάκτησης κυρίαρχης θέσης στην αγορά από οποιαδήποτε εταιρεία και εφόσον πρόκειται για συμπεριφορά ενάντια του ανταγωνισμού, και έχουμε παραδείγματα και μάλιστα η Κομισιόν τακτικά ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις, τότε θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά μέτρα. Γιατί και εδώ υπάρχει ένας τρόπος, κρύβεται ένας τρόπος ομοιομορφίας για το περιεχόμενο. Θα υποβάλω λοιπόν ε, τέτοιες τροπολογίες για να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση και ελπίζω να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο εργασίας για το οποίο και σας ευχαριστώ. Και τώρα, να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ορίζεται την 9η Φεβρουαρίου. Θέλετε να έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες και όλους για τα πολύ χρήσιμα σχόλια. Θα ήθελα πρώτα να καθησυχάσω τα πρόσωπα εκείνα που εξέφρασαν ανησυχίες. Δεν νομίζω ότι εμποδίζοντας τον γεωγραφικό αποκλεισμό μειώνεται την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην πρότασή μου. Επιθυμώ να διασφαλίσω ότι όλο το περιεχόμενο το οποίο παράγουν οι παραγωγοί, οι συγγραφείς μας κλπ. να μπορεί να διαδίδεται όσο γίνεται ευρύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αμείβονται για το έργο τους. Κάθε ένας που επιτρέπει να διαδίδεται το έργο του θα πρέπει αυτό να γίνει διάδοση, δηλαδή αυτή να γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν τις συγκεκριμένες άδειες. Αυτό θα εξυπηρετήσει και θα ωφελήσει ιδίω τις μικρές χώρες Αναρωτηθείτε, πόσες φιλανδικές ταινίες έχετε δει ή γνωρίζετε την ύπαρξή τους. Σουηδικές, Πορτογαλικές, Πολωνικές. Ίσως μερικές από τις ε, ταινίες αυτές να έχουν ε, προωθηθεί πολύ καλά στην χώρα τους, αλλά μετά να έχει πέσει η λεπίδα του γεωγραφικού αποκλεισμού και να μην προχωρούν σε άλλες χώρες. Ας φροντίσουμε λοιπόν έτσι να διευρυνθεί το ακροατήριο που τις παρακολουθεί, το κοινό. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για κλοπή της διανοητικής ιδιοκτησίας ορισμένων δημιουργών. Αντίθετα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διευρύνουμε το πεδίο διάδοση των έργων τους. Θα εξυπηρετήσει η ποικιλία αυτή, η πολυφωνία αυτή. Και ο έλεγχος θα είναι καλύτερος και πιο αποτελεσματικός. Θα πρέπει να ομολογήσετε ότι Η αμερικανική κουλτούρα, ιδιαίτερα στου τομεί αυτού, επειδή είναι απολύτω ελεύθερη από γεωγραφικού αποκλεισμού, έχει γίνει και η κυρίαρχη στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πάντοτε μέσα στα πλαίσια τη νομιμότητα. Και βεβαίω να, να είμαστε εξοπλισμένοι με τι αναγκαίε άδειε. Συμπεραίνοντα, η πρότασή μου θεωρώ ότι δεν κρύβει κινδύνου, ιδίω ό,τι αφορά περιεχόμενο που υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματική διοκτησίας. Για τι τιμέ τώρα των διαφόρων ψηφιακών υπηρεσιών. Α πάρουμε το Netflix ω παράδειγμα. Το οποίο πωλεί τις υπηρεσίες του σε διάφορε χώρε. Και είναι αληθέ ότι είναι διαφορετικό ο λογαριασμό που πληρώνεται τελικά ανάλογα με τον τόπο που βρίσκεστε. Αν η προσφορά υπηρεσιών είναι πιο περιορισμένη, πληρώνεται λιγότερα και ούτω καθεξής. Καλό παράδειγμα αυτό για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, διότι δεν είναι κατάλληλη λύση. Ας πάρουμε τα τέλη περιαγωγής. Θυμούμε όταν πρώτο ήρθα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προ 13 ετών, τα τέλη περιαγωγής ήταν διαφορετικά από χώρα σε χώρα, με πολύ διαφορετικές βασικές αρχές. Ακόμη και αν καλούσατε κάποιον και ε, δεν απαντούσε. Παρ' όλα αυτά ε, σας καλούσαν να πληρώσετε πολλά χρήματα. Αυτά τα καταργήσαμε. Ίσως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Εάν μπορεί κανείς να αυξήσει τους αριθμούς των πελατών, τότε οι τιμές θα πέσουν. Το κάναμε αυτό με την περιαγωγή. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο τώρα και με την αποφυγή του αποκλεισμού ανάλογα με την κατοικία του καθενό. Και συμφωνώ με την κυρία Ρέντα, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων, αν εξετάσετε τι προτάσει που ήδη έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν εγκριθεί από εμά, θα δείτε ότι έχουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μπορούμε να ε, θεσπίσουμε. Δεν κάνουμε κανένα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε το άλμα και βεβαίως προηγείται η ανάλυση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει εάν αφαιρέσουμε τον γεωγραφικό αποκλεισμό για ορισμένα έργα τα οποία προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθούμε από την προσπάθεια. Συν το χρόνο θα καταλήξουμε σε μια επαρκή λύση. Έχοντας παρακολουθήσει την συζήτηση, και ακούσει τα σχόλιά σα, αναμένω τη συνεργασία μαζί σας και είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε εν τέλει να συντάξουμε ένα έγγραφο το οποίο θα γίνει δεκτό από την Επιτροπή Προστασία Καταναλωτών που αυτή ω γνωρίζετε είναι αρμόδια επί και αυτό που θέλω να διασφαλίσω είναι ότι η δική μα γνωμοδότηση θα περιλαμβάνει τι αναγκαίε νομικές διατάξεις ώστε να επιτρέψει στην πρόταση να λειτουργήσει πράγματι υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση του θέματος αυτού και συνεχίζουμε με το υπαριθμό 27. Εξέταση γνωμοδότησης για την απόσπαση εργαζομένων στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών. Το λόγο είχε ο κύριος Καβαντά. Merci, Président, chers collègues. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Για την σύνταξη της γνωμοδοτήσεως έλαβα υπόψη την θαυμάσια γνωμοδότηση που μας κοινοποιήθηκε από την νομική υπηρεσία για να μπορέσω να συγκεντρώσω την προσοχή μου, ειδικά στις αρμοδιότητες βέβαια της Επιτροπής μας. Οι κανονισμοί είναι Ρώμη 1 και Βρυξέλλες 1 με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τα άλλα ε, νομοθετικά εργαλεία σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμεθοριακά από αποσπασμένους εργαζομένους και σε ό,τι αφορά την συμβατότητα ορισμένων πτυχών της προτάσεως με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Επ' αυτού συνέταξα γνωμοδότηση ιδίως προτείνοντας νέους μηχανισμούς και ενισχύοντας τους υφιστάμενους για να διευκολυνθεί η παροχή διαμεθοριακά υπηρεσιών, προσπαθώντας βέβαια να προλάβω καταστρατηγήσεις, απάτες και ούτω καθεξής. Πρόσεξα ιδιαίτερα την κοινωνική προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων, διότι πρόκειται για κατηγορική επιταγή για να εξασφαλιστεί η κοινωνική αρμονία στην Ευρώπη και υποστηρίζω ιδίω την αρχή της ισότητας μεταχείρισης και την αποφυγή οποιασδήποτε, αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης, οποιασδήποτε διάκρισης στη βάση εθνικότητας. Ο κανονισμός Ρώμη 1 επιτρέπει με γενικό τρόπο στους εργαζομένους και εργοδότες να εφαρμόζουν το εργατικό δίκαιο χωρίς να στερείται ο εργαζόμενος την προστασία του δικαίου που του εξασφαλίζει την ευνοϊκότερη μεταχείριση ή, εν πάση περιπτώσει, στην βάση του οποίου, ή μάλλον η, χώρα, της χώρας δηλαδή, όπου ε, ε, επιτελεί το έργο του βάζω μια περίοδο 24 μηνών από την οποία και μετά η χώρα υποδοχής θεωρείται η χώρα στην οποία κατά συνήθιν απασχόληση εργάζεται ο εργαζόμενος. Αυτό βέβαια είναι ειδικό κανόνας που αποκλίνει από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού Ρώμη 1, όμως είναι σύμφωνο με τον προσωρινό χαρακτήρα της αποσπάσεως και επομένως τα, τα δύο, ε, οι δύο αυτοί μηχανισμοί δεν είναι, δεν είναι αλληλοποκλείονται, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτή η πρόταση αναθεωρήσεως θεωρήθηκε από ορισμένου ως περιορισμός της ελευθερίας προσφοράς υπηρεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης. Ωστόσο, το δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι η κοινωνική προστασία των εργαζομένων αποτελεί αποχρόντα λόγο και ο περιορισμός των 24 μηνών είναι απολύτως δικαιολογημένος και δεν αντιβαίνει στην αρχή ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, επιτρέπει αντίθετα την βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων. Άλλο σημαντικό θέμα της νομοδοτήσεως είναι ότι τονίζει τον προβληματισμό της διπλής απόσπασης των προσωρινά, προσωρινά εργαζομένων, προσωρινά εργαζόμενων μισθωτών. Πράγματι, με την αύξηση του αριθμού των προσωρινά εργαζόμενων, μειώνονται οι έλεγχοι και μειώνονται οι ευθύνες. Εν τέλει, η διάθεση εργαζομένου από μια επιχείρηση ευρέσεως εργασίας σε χώρα μέλος, σε μια χώρα μέλος της οποίας είναι, έχει την υπηκότητα ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να θεωρηθεί απόσπαση. Εκτός εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως συνήθις διαμονή, διαφορετική συνήθις διαμονή, εάν αυτή αιτιολογεί τέτοιο χαρακτηρισμό για να αποφευθούν απάτες που γνωρίζετε και που είναι συνήθις στην αγορά εργασίας για την εξασφάλιση της απασχόλησης του αποσπασμένου εργαζόμενου και για την αντιμετώπιση επιχειρήσεων που είναι εικονικές, θεωρώ ότι η επιχείρηση η οποία αποσπά εργαζόμενο σε μια άλλη χώρα μέλος, σε άλλη χώρα μέλος βεβαίως, θα πρέπει να μπορεί όχι μόνο να αιτιολογεί την ύπαρξη έδρας σε αυτή την άλλη χώρα, αλλά και να διασφαλίζει ότι ο κύκλος εργασιών της όντως υλοποιείται στη χώρα μέλος όπου έχει την έδρα της. Άρα ότι δεν ε, είναι φτιασιδωμένη η επιχείρηση. Στην βάση δηλαδή αυτή. Εγώ προσέχω ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Πρόκειται για ένα θέμα καυτό για όλες τις χώρες μέλη συζητήθηκε και πάρα πολύ στην προεκλογική εκστρατεία, το είδαμε αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία, το ακούμε βεβαίω να συζητείται και στην Ολλανδία αλλά και στην Γαλλία, ε, συζητείται πολύ και στη Γερμανία, άρα θα προσέξω πάρα πολύ τα σχόλια που θα μου υποβάλλετε και πρέπει οπωσδήποτε να μπει τάξη σε αυτή την αταξία η οποία υφίσταται σήμερα. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους τους συναδέλφους. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Εσείς κύριε Σάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Καβαδά για την έκθεσή του. Να μου επιτρέψετε να κάνω δύο σχόλια. Ένα κάπως περισσότερο πολιτικό και το άλλο έχει νομικό χαρακτήρα. Το πολιτικό σχόλιο έχει την έννοια διευκρίνησης ο κανονισμός αποσπάσεως εργαζομένων είναι παλαιότερος από την μεγάλη ενοποίηση της Ευρώπης τότε, το 2004 και βέβαια το 2012 που μπήκαν και άλλες ε, ανατολικές χώρες στην Ευρώπη. Πολύ σοφά δεν θεώρησε τότε η Ευρώπη ότι θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτή τη λύση αν και, υπάρχουν, και υπήρχαν μεγάλες αποκλήσεις με, μεταξύ των χωρών με τη μεγάλη αυτή διεύρυνση. Τώρα όμως που έχουν περάσει 10 ε, χρόνια και περισσότερα βλέπουμε ότι δεν μειώθηκαν πραγματικά οι αποκλήσεις τουλάχιστον όχι στο βαθμό που ελπίζαμε όταν ενταχθήκαμε το 2004. Τώρα, ο κανονισμός αυτός που έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και η βασική μου ανησυχία και στις προηγούμενες συζητήσεις ήταν ότι πάμε να αναθεωρήσουμε κάτι το οποίο άπτεται της κοινωνικής πολιτικής και για προφανείς λόγους διότι σε δυτικές ευρωπαϊκές χώρες το κοινό αντιλαμβάνεται την απόσπαση εργαζομένων αλλά και την διακίνηση, την ελευθερία διακίνησης εργατικού δυναμικού ως κάτι το οποίο ε, είναι επιζήμιο για την ε, κοινωνική δικαιοσύνη στις χώρες τους, για τους μισθούς κτλ. Έχουμε και την οδηγία περί που έχει ξεσηκώσει ορισμένα συνδικάτα στην Ευρώπη και υπήρξε αντίσταση κατά της ελευθερίας διακινήσεως εν τέλει. Αυτό είναι και το πλαίσιο με στο οποίο συζητούμε τώρα. Κατανοώ απολύτως. Βεβαίως, οι του κοινού είναι σημαντικές. Αυτό που αντιλαμβάνεται το κοινό, δηλαδή ως κάτι ανησυχητικό, έστω και αν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά πάντως οι ανησυχίες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται. Εγώ θεωρώ, και έρχομαι τώρα στο νομικό επιχείρημα, Θεωρώ ότι η επιλογή της οδηγίας, μάλλον με την οδηγία, θα τροποποιήσουμε κάποιους βασικούς κανονισμούς και εν προκειμένου τον κανονισμό Ρώμη 1. Αλλά αυτή δεν είναι η σωστή νομική επιλογή κατά τη γνώμη μου. Επιμένω ότι κατανοώ ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Υπάρχουν όμως και κάποιες αρχές που είναι η αρχή προσφοράς υπηρεσιών. Είναι η αρχή της διακίνησης του εργατικού δυναμικού, της ελευθερίας δηλαδή διακίνηση των εργαζόμενων. Αυτές είναι αρχές που μας στηρίζουν ακόμα και σε δύσκολου καιρού. Εγώ θεωρώ τον κανονισμό και ιδίω εκείνη την μαγική φόρμουλα ότι ε, η απόσπαση μετά από 24 μήνες πάβει να είναι απόσπαση, το θεωρώ ως κάτι που δεν είναι σωστά διαθρωμένο, διότι εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε κάποιους κανονισμούς, θα πρέπει εκεί να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή στον Ρώμη 1 και όχι θεσπίζοντας κάτι το οποίο προκαλεί ε, ανασφάλεια δικαίου. Έχουμε και την ε, γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας, η οποία ε, λαμβάνει κάποιες θέσεις. Εν των θέσεων της νομικής υπηρεσίας από αυτού, για, το, για τα πολύ σημαντικά ερωτήματα που τους θέτουμε να μας δώσουν νομικές διευκρινήσεις, μας υποβάλλουν απόψεις με χαρακτηρισμούς όπως αναλογικό ή αιτιολογημένο. Όμως, άλλοι νομομαθείς λένε άλλα πράγματα και οι δικαστές όταν εξετάζουν τα στοιχεία θεωρούν ότι αυτά δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν είναι conclusive δηλαδή. Ακούμε δηλαδή οι νομικές γνώμες για μένα η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας είναι σαφής ότι αυτός ο κανονισμός αντιτίθεται στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Αλλά είναι, λέει, αιτιολογημένος και είναι και αναλογικός. Αυτό είναι το συμπεράσμα του. Από τη σκοπία, τη δική μου όμως, αυτό δεν είναι το θέμα. Ότι ο κανονισμός ή τέλο πάντων η τροποποίηση του κανονισμού είναι αντίθετη με την ε, ελευθερία παροχής υπηρεσιών. είτε είναι αναλογικό, είτε είναι αιτιολογημένο. Αυτό παραμένει ως ερώτημα και μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο και όχι βέβαια μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο κατανοώ ότι υπάρχουν διαφορές θέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν όμως επιχειρήματα και στην έκθεση του κ. Καβαντά αλλά και στην αιτιολόγηση των αλλαγών των τροποποιήσεων δηλαδή, που φαίνεται να δείχνουν ότι όταν μιλούμε για κοινωνική προστασία εργαζομένων, δεν θα πρέπει να εξετάζουμε μόνο την κοινωνική προστασία εργαζομένων στο ένα μέρο τη Ευρώπη, αλλά και στο άλλο. Τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται και κυρίω από κεντρικέ και ανατολικέ χώρε τη Ευρώπη, αυτοί που εργάζονται εκεί και αυτοί έχουν ανάγκη κοινωνική προστασία να διατηρήσουν δηλαδή τις δουλειέ τους διότι αλλιώς δεν θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ούτω καθεξής. Εξακολουθώ να βλέπω λοιπόν αυτή την διαίρεση Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Και ο κανονισμός δεν αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Όμως, έρχομαι στο συμπέρασμά μου. Εμείς είμαστε Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Δηλαδή, καλούμεθα να εξετάσουμε το θέμα. Κοιτάξτε, ε, Επιτροπή Απασχολήσεως και λοιπά εξετάζουν την ευρύτερη οπτική. Αυτό που οφείλουμε να εξετάσουμε εμείς είναι αν ο κανονισμός που επιλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν ο τρόπος που επιλέγει να αντιμετωπίσει το κοινωνικό αυτό πρόβλημα είναι σωστός ή όχι. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι, διότι αντιβαίνει στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών. διότι η επιλογή των 24 μηνών είτε είναι κατ' επιλογή, είτε είναι υποχρεωτικός κανόνας, παρόλα αυτά εμποδίζει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Και τι να το κάνουμε αυτό. Γιατί να επιλέξουμε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι δικαιολογημένο, αιτιολογημένο αν θέλετε και αναλογικό. Έχω και μια διαδικαστική ερώτηση. Η Επιτροπή Απασχολήσεως έχει κάνει κάποια προσαρμογή και έχει αναβάλει την ημερομηνία τους, τη δική τους δηλαδή, κατά θέσεω τροπολογιών. Θα ήθελα λοιπόν αναλόγως να τροποποιηθεί και η δική μας. Ευχαριστώ. As well, uh, Joseph, do you have an idea? Ευχαριστώ. Έχετε μια ιδέα μέχρι πότε θέλετε να αναβληθεί η προθεσμία. I am not technician on that. Όχι. Ε, ξέρω ότι η Επιτροπή Απασχόλησης το έχει αναβάλει μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω όμως ακριβώς πότε είναι οι συνεδριάσεις τους. Ε, απλώς χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο από τις λίγες μέρες που έχουμε τώρα. Ε, okay, Mr. Voss. Vielen Dank. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω τόσο είπε ο κύριο Σάιερ έχω την αίσθηση ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να μελετηθούν περισσότερο. Τρία συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο ίσως έχει και κάποιο πολιτικό εκτός από το νομικό χαρακτήρα. Στον κανονισμό Ρώμη 1, εξ όσων καταλαβαίνω, έχουμε την ελευθερία επιλογής, μια συμβατική ελευθερία δηλαδή, που κατά τη γνώμη μου, περιορίζεται χρονικά στους 24 μήνες τώρα με την πρότασή σας. Αυτό μου φαίνεται κάπως αυθαίρετο, γιατί έχει πέντε χρόνια. Γιατί δύο χρόνια. Ίσως μετά να γίνει μονάχα ένας χρόνος ή μόνο έξι μήνες. Για να καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο συμπέρασμα. Τα οποία νομικά ίσως να έχουν καλώς, αλλά πάντως εδώ βρίσκω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι πάντοτε είμαστε υπέρ της συμβατική ελευθερίας, της ελευθερίας των συμβάσεων δηλαδή. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε. Εξάλλου διαρωτώμε με θα είναι οι επιπτώσεις. Εάν όντως επιλέξουμε τους 24 μήνες, εάν εγώ ως Γερμανός αποσπώμαι στο Βέλγιο και μετά από 24 μήνες υπόκειμαι απολύτως στο βελγικό δίκαιο, αλλά έχω μια διαφορά με τον εργοδότη μου στην Γερμανία αυτό, από ό,τι κατανοώ εγώ, θα οδηγήσει στο ότι τα γερμανικά δικαστήρια θα κληθούν να ελέγξουν το βελγικό δίκαιο. Δεν είμαι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο πραγματικά εξυπηρετεί. Ή αν ίσως προκαλεί υπερβολικές περιπλοκές στην υπόθεση. Μήπως είναι σωστό να σκεφτούμε εάν όντως θα είναι αυτές οι επιπτώσεις από τον, από τον κανόνα αυτών, δηλαδή ότι πλέον τα εθνικά δικαστήρια θα έρχονται να εγκύψουν στο εθνικό δίκαιο άλλων χωρών μελών. Κάτι που νομίζω ότι οδηγεί σε μια αφόρητη περιπλοκότητα της ε, ρύθμισης. Ένα άλλο που ίσως είναι περισσότερο ένα πρόβλημα που απορρέει από το γερμανικό δίκαιο, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλες χώρες μέλη, η ελευθερία συλλογικών συμβάσεων που περιλαμβάνεται στο άθρο 9 του Γερμανικού Συντάγματος και η ελευθερία των συλλογικών συμβάσεων σημαίνει επίσης ότι έχω το δικαίωμα και να μην συμμετάσχω. Δηλαδή δεν θέλω να υπάρξει τώρα όμως μια αρνητική ελευθερία με την έννοια ότι δεν συμμετέχω. Εάν τώρα αυτή η ρύθμιση επιβληθεί στο δηλαδή δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων, τότε μπορεί να οδηγήσει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανταγωνισμού στο νομικό αυτό τομέα. Αυτό δηλαδή, κάτι δηλαδή το οποίο είναι συνταγματική επιταγή στην Γερμανία, το δικαίωμα δηλαδή να πει κάποιο ότι δεν θέλω συλλογική σύμβαση, μπορεί να είναι υποχρεωμένο όμω από το ευρωπαϊκό δίκαιο να τη δεχτεί. Εδώ χρειάζεται κάποια λύση, διότι αλλιώ το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει και μέσα στην δογματική ανατένιση του δικαίου. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύσεις και επειδή ακριβώς είναι τόσο περίπλοκο νομικά θα προτείνω όντως να δοθεί μια αναβολή για να έχουμε τη δυνατότητα να εγκύψουμε σε λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Εσείς κύριε είναι. Εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και να πω ότι με την πρώτη μονάγνωση της πρότασης ε, φαίνεται να είναι πολύ καλή. Πρόκειται για μια πρόταση που στόχο έχει να ενισχύσει αυτό που περιγράφει ενώ προστατεύει με την ελευθερία κυκλοφορία θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε ο κόσμο να έχει ευκαιρίε, να έχει ευκαιρίες, αλλά όχι για να διευκολύνουμε την κατάχρηση και τι διακρίσει. Γι' αυτό και συμφωνώ με τι ε, βασικέ γραμμέ τη πρόταση. While fixing the real problems that we have with discrimination today, να τονίσουμε και να διευρύνουμε ε, τις κανόνες κατά των διακρίσεων, αλλά χωρίς να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα, όπως ας πούμε συγκεκριμένα ότι οι λύσεις που στηρίζουμε δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα για τους το δικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων που λειτουργεί ε, καλά, αλλά ε, σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν προβληματικέ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα το προσέξω πάρα πολύ. Και επίσης η ιδέα για ίση πληρωμή όλων των εργαζομένων για την ίδια δουλειά ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί. Βλέπω την ώρα και είμαι πεπισμένο εξάλλου πώ θα ξαναπανέλθουμε σε αυτό το θέμα επαναλημμένα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, κυρία Ρέγκναρ. Ευχαριστώ και εγώ βέβαια κοιτάζω το ρολόι και γι' αυτό θα συντομεύω πρώτον. Λυπούμε που η κυρία Ντελβό δεν είναι, που είναι η συγκρότηση, μας δηλαδή, δεν είναι παρούσα, δεν είχε αντιληφθεί ότι το ζήτημα Α, να τη, να τη. Ελπίζω ότι θα λάβει το λόγο. Ε, έτσι εγώ λοιπόν θα είμαι σύντομη. Η συμβατότητα με τον ε, κανονισμό Ρώμη 1 είναι δεδομένη. Αυτή είναι η άποψή μας. Και για το επιχείρημα του κυρίου Βόση για τους 24 μήνες, αυτό ανταποκρίνεται και στο streamlining του ε, κανονισμού 883. Για το συνολικό πλαίσιο βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε πραγματικά στην καρδιά, στον πυρήνα των πολιτικών θεμάτων που ε, συζητούμε σήμερα έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι για όλους και όλους μας εδώ στόχος είναι οι μεγάλες μισθολογικές και κοινωνικές διαφορές να μην μεγαλώσουν κι άλλο, αλλά αντίθετα να προσεγγίσουμε οι μεν τους δε και επομένως με κάθε νομικό μέσο που διαθέτουμε και που εγκρίνουμε εδώ να φροντίσουμε να προχωρήσουμε σε μια προσέγγιση και όχι σε μια απόκληση που δυστυχώς τη βλέπουμε. Γι' αυτό και εδώ στην Νομική Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουμε τα προβλήματα αυτά μέσα από αυτή τη γωνία. Ως Αυστριακή δεν μένω αδιάφορη όταν εργαζόμενοι σε αυστριακές επιχειρήσεις γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση επειδή προέρχονται από την Αλοδαπή Είναι αυτές ακριβώς οι κοινωνικές ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με στόχο να συμφωνήσουμε σε ελάχιστα πρότυπα. Και επειδή τώρα βέβαια έρχεται και η ώρα της ψηφοφορίας θα αρκεστώ μόνο σε αυτά. Αλλά αυτό είναι το νόημα νομίζω της εργασίας της Νομικής Επιτροπής. Εσείς κύριε Βόση. Ευχαριστώ πολύ σύντομα να απαντήσω στην κυρία Ρέγνερ η οδηγία 883 δίνει τη δυνατότητα να υπερβεί κανείς και το όριο των 24 μηνών και στην πράξη μέχρι 5 έτη. Ας το σκεφτούμε και αυτό λοιπόν, εάν δηλαδή θέλουμε ευθυγράμμιση. Αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η απάντησή μου. Το άρθρο 16 της εν λόγω οδηγίας δίνει τη δυνατότητα να ε, υπερβείτε το όριο των 24 μηνών. πληροφορήθηκα ότι η αρμόδια επιστουσία η Επιτροπή Απασχολήσεως θα ψηφίσει την έκθεσή της τον Ιούνιο. Ακόμα περισσότερο, τον Ιούλιο, δηλαδή 7ο μήνα. Άρα έχουμε αρκετό χρόνο και ίσως μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτούς ένα μήνα ακόμη, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Δεν θα πρέπει νομίζω να είναι πρόβλημα αυτό. Ας πούμε λοιπόν 28 Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου. Ε, έχει όντως 28 φέτος ημέρες ο Φεβρουάριος. Άρα, ε, λίγη εδώ η συζήτηση του θέματος για την ώρα. Εσείς Ζλωτόσκι, ορίστε. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Λίγα λόγια. Για το ίδιο θέμα. Βεβαίως και υποστηρίζω το αίτημα του κ. Σάιερ να παραταθεί δηλαδή η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Επιτρέψτε μου όμως να πω λίγα λόγια ακόμη για τις προτινόμενες αλλαγές. Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προκαλεί ορισμένα ερωτηματικά σε ό,τι αφορά θεμελιώδη νομικά θέματα περιορισμός δηλαδή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών εν τέλει. Και εν τέλει χρειάζεται να δοθούν εγγύησεις και σε εργοδότες και σε εργαζόμενους. Η νομική γνωμοδότηση που ζήτησε η Επιτροπή μας ομολογώ δυστυχώς ότι δεν κατόρθωσε να άρει όλες τις αμφιβολίες που είχα και ιδίως ό,τι αφορά τον κανονισμό Ρώμη 1 και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη δε τροπολογία υπαριθμών 3 ο ΣΥγητή προσπαθεί να απαλύνει τις ε, αμφιβολίες αυτές. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Η προσπάθεια δεν είναι αρκετή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το μείγμα αυτό των αλληλοσπαρασόμενων κανονισμών, των αλληλοσπαρασόμενων διατάξεων σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο οι διαφορετικές νομοθεσίες εργατικού δικαίου αν έχετε μία εταιρεία και διαφορετικές χώρες όπου αποσπώνται εργαζόμενοι θα σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούνται πολύ διαφορετικά συστήματα και ταυτόχρονα θα είναι και βαρύτατο το γραφειοκρατικό άκθος. Επίσης η μείωση στους 24 μήνες θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα είναι αδύνατο να λειτουργήσουν πολλές επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Θα είναι πολύ δύσκολο να θεμελιωθεί αυτό. Ιδίω εφόσον οι συνθήκες μας δεν προβλέπουν τέτοιες, τέτοιους περιορισμούς. Δεν δικαιολογείται λοιπόν επιβολή τέτοιου περιορισμού, ιδίω σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Η δε τροπολογία 5 επίσης δεν απαλύνει τις αμφιβολίες μου. Ίση μεταχείριση για αποσπασμένους και ντόπιου εργαζόμενου, δεν θα πρέπει να οδηγήσει, να οδηγήσει σε διακρίσει σε βάρος των αποσπασμένων εργαζομένων που θα στερούνται πολλών ε, ωφελημάτων, για παράδειγμα την ε, κάλυψη των εξόδων διαμονής τους. Τα δε επιχειρήματα της νομικής υπηρεσίας που λένε ότι γραφεία ευρέσεως εργασίας θα μπορούν να απασχολούν ανθρώπους μόνο για περιορισμένο διάστημα αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας του 2008 για την ε, προσωρινή απασχόληση. Λέει ότι εκεί, ότι οι προσωρινά εργαζόμενοι μπορούν να απασχολούνται και με ε, ε, συνήθεις συμβάσεις εργασίας. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός μεταξύ των χωρών μελών. Ιδίως στον αγώνα κατά των άδικων πρακτικών. Είναι δύσκολο όμως να συμφωνήσει κανείς με τον εισηγητή, ο οποίος λέει στο τέλος του κειμένου του ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βαίνει στην σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά των καταχρήσεων. Εγώ νομίζω ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως μάλιστα επιδεινώνει τα προβλήματα και ιδίως σε ό,τι αφορά το κόστος, το διοικητικό κόστος ε, των νομικών υπηρεσιών και που εν τέλει μπορεί να, μπορούμε να δούμε, να δούμε να μειώνονται οι αριθμοί αποσπασμένων εργαζομένων στην Ευρώπη. Οι προτινόμενες αλλαγές αποτελούν διακρίσεις σε βάρος αποσπασμένων εργαζομένων από τις νέες χώρες μέλη. Αν αυτό είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε τον έχει επιτύχει. Όμως θα είναι πολύ δύσκολο να εγκριθεί ή να θεωρηθεί ότι είναι επαρκής αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ σύντομα τώρα πια ο κύριος Καβαντά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Συνειδητοποιώ ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που θίγει συμφέροντα, τα οποία βλέπουμε να διαμορφώνονται εδώ και μία δεκαετία. Είναι ένα θέμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα στον κόσμο της εργασίας και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις συζητήσεις μας. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω με την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στο θέμα και να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία ως έχει δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση τώρα. Θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες.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 Uh, Μου ζητήθηκε από τη Γραμματεία να ετοιμάσετε τις κάρτες σας έτοιμες, γιατί σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ακόμα και οι γνωμοδοτήσεις θα ψηφίζονται με ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο θέμα που έχουμε να ψηφίσουμε είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Χρυσόγονου Οδηγία 2004-37, κάθετο 37. Λοιπόν, τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 49, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 49. Μάλλον έγινε δεκτή, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Ναι, πράγματι. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή μάλλον, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την ενεα. Απερίφη. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 12. Απερίφθη. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ όχι 29 έχει καταπέσει συμβιβαστική 1 υπέρ δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική οκτώ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τέλος το απολογημένο ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Εκτή συγχαρητήρια προς τον κύριο Χρυσόγωνο. Έχουμε τώρα δύο συγκεκριμένες ψηφοφορίες, η μία σχετικά με την έκθεση Κοφεράτη 36 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την έκθεση Κοφεράτη. Συγχαρητήρια στον κύριο Κοφεράτη, δεκτή. Η επομένη είναι η έκθεση της κυρίας Μπουτονέ. Ψηφίζουμε. Κοιτάξτε, αναφέρομαι στο σημείο 17, η έκθεση της κυρίας Μπουτονέ. Μοναδική ψήφος. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε για μια ακόμη φορά. για το σημείο 17 ηλεκτρονική ψηφοφορία Τέλος της ψηφοφορίας έγινε δεκτή συγχαρητήρια στην κυρία Μπουτονέ. Το σημείο 18. Πάντα έκθεση μπουτονέ, ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια στην κυρία Μπουτονέ. Σημείο 19. Έκθεση Καβαντά. Συγχαρητήρια στον κύριο Καβαντά. Και τώρα έχουμε την απαλλαγή του προϋπολογισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 και 4 υπέρ, α, συγγνώμη, έχουν καταπέσει αυτές. 3 υπέρ, Α, έχει καταπέσει και αυτή η διορθώνη ο πρόεδρος. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή εννέα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την εννέα παρακαλώ. Δεκτή. έντεκα υπέρ Α, όχι, η 11 έχει καταπέσει, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης ψηφίζεται. Για... Λείπει μία ψήφος. Τέλος λοιπόν της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή η πρόταση. Συγχαρητήρια στον κύριο Λεμπρετό. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τους συντονιστές. Yeah.